ήταν στο Γαλλικό Κοινοβούλιο και έτσι λοιπόν διαπιστώνεται η χειρία των θέσεων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 19 Ιουνίου 2017. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής ε, Δημοκρατίας ε, ανακοίνωσαν στον Πρόεδρο την εκλογή της κυρίας Κριστέλ Λεσεβαλιέ και της κυρίας Μαρή Πιέρ Η κυρία Λεσεβαλιέ και η κυρία Διού αντικαθιστούν την ε, κυρία Μαρή Λεπέν και τον κύριο Μελάνσου, από 19 Ιουνίου 2017. Σας καλωσορίζω συνάδελφοι και να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Λεζεβαλιέ και η κυρία Βιού ε, έχουν πλήρη δικαιώματα για τη συμμετοχή